έχω από το ΕΛΚ, ECR, Πρασίνους και ΕΝΕΛ, αιτήσεις τροποποιήσεων ως προς τους διορισμούς που θα εγγραφούν στα πρακτικά. Εάν δεν θα υπάρξουν παρατηρήσεις στα πρακτικά, τότε θα επιβεβαιωθούν